and it's late, Chairman, and it's unacceptable. Okay. Then, uh, Vox Populi, so... Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αφού αυτό απαιτεί ο λαός. Όχι, να μην ξεκινήσουμε. Yes. That, I think. Our chairman is coming in few minutes. Σε μερικά λεπτά θα είναι εδώ και ο πρόεδρός μας. Μπορείτε να ξεκινήσετε κύριε Πρόεδρε και μετά να δώσετε την Προεδρία στον Πρόεδρο όταν εμφανιστεί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ψηφοφορία. Απαλλαγή 2012, Γενικός Προϋπολογισμός, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η εισηγήτρια κυρία Μαρία Μουνίθ. Θέλετε να πάρετε το λόγο, όχι. Πολύ ωραία. Συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Μάλλον όχι. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Μάλλον όχι, λέει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να πάμε στην τροπολογία 7.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 Πέρα τη ψηφοφορία 37 ψήφοι υπέρ, 39 μάλλον, γιατί έχουμε δύο συναδέλφους χωρίς ε, τις κάρτες τους, τρεις ε, ψήφοι κατά, τέσσερις αποχές, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια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 τον αρμόδιο Υπουργό για τα θέματα τα ευρωπαϊκά της Ουκρανίας και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να καθυστερήσω και με την, και με την κυρία Άστον. Ερχόμαστε λοιπόν για, τον, ε, ε, για την απαλλαγή τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ <clears throat> κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές και πάλι. 8 κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, ε, καμία ψήφος κατά και 5 αποχές εγκρίνεται. Τώρα, ε, σχέδιο σύσταση προς το Συμβούλιο. Κύριε Βότσον, έχετε το λόγο. Σερ Γκράμ, έχετε το λόγο. Μήπως μπορώ να κάνω μία αίτηση προς ε, εμάς. Μετά από τη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, <clears throat> θέλουμε να αλλάξουμε τον τίτλο της έκθεσης. Σύσταση για τη χρήση τηλεοπτικών, ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην στην ευρωπαϊκή διπλωματία και όχι σαν εργαλείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Και η συνέλευση των Πρόεδρων νομίζω ότι συμφωνεί. Απλώς χρειάζεται να υπάρξει μια επίσημη αίτηση από την Επιτροπή μας και νομίζω ότι υπάρχει η υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι γιατί έχει υποδειχθεί σωστά ότι αν αναφερθεί ως εργαλείο της ευρωπαϊκής διπλωματίας είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε προπαγάνδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Και κάποια μέλη, ιδίως το ΕΛΚ, η κυρία Πακ και άλλοι, ε, ήταν κατά της έκθεσης να καθυστερήσουν κατά τι συγγνώμη, να καθυστερήσουν την έκθεση για αυτό το λόγο. Εγώ σας παρατρύνω να μην την καθυστερήσουμε. Κάναμε τι απαραίτητε συζητήσεις στην Επιτροπή μας, συναντηθήκαν και οι και νομίζω <clears throat> ότι μπορεί να εγκριθεί αυτή η σύσταση ώστε να έρθει στην Ολομέλεια, τον, ε, στην ε, Ολομέλεια 2 του Φεβρουαρίου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την υποστήριξη που μου δώσαν σε αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε σήμερα. Ακόμα και αν αλλάξει ο τύπος, ακόμα υπάρχει κάτι το παραπλανητικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε μια τέτοια έκθεση που θέλουμε να εγκρίνουμε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία είναι πλήρης παρανοήσεων. Οποιοδήποτε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να μας κατηγορήσει ότι θέλουμε να κάνουμε προπαγάνδα ως Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Euronews και άλλων τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό είναι ουσιαστικά κάτι το πολύτιμο για τους εχθρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Ένα παράδειγμα σας πω. Έχουμε μια συμβαστική λύση όπου κανονικά δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Λέει να δημιουργήσουμε μια χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ραδιοτηλεοπτικά, τονίζοντας τις αξίες για τη ραδιοτηλεόραση και προωθώντας την αντικειμενικότητα της, των εκπομπών κτλ. Μα ποιος θα το κάνει αυτό. Όλα αυτά είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο ξεκινάει από ευσεβείς πόθους και καλές ε, θελήσεις, αλλά όλα αυτά θα είναι <clears throat> όπλα εναντίον μας από τους εχθρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε τι θα πει ο κύριος Φάρας και το UKIP εναντίον όλων αυτών. Σας παρακαλώ λοιπόν αυτή την έκθεση να την απορρίψουμε και ή αλλιώς να ψηφίσουμε εναντίον. Γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό κάνουμε ένα λάθος, κάνουμε ένα αυτογκόλ σε βάρο μας. Εγώ δεν ήξερα ότι θα ερχόταν αυτή η έκθεση στην ημερήσια διάταξη και η Επιτροπή μας δεν είχε επιληφθεί για το θέμα αυτό γιατί αλλιώς θα είχαμε παρέμβει νωρίτερα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά ποτέ δεν είναι αργά για να σταματήσουμε κάτι το οποίο θα μας βλάψει όλους απαξάπαντες. Διαβάστε το κείμενο, θα είναι σε βάρος μας όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι και εγώ έμαθα τη θέση της συναδέλφου Ντόρις Πάκ μετά από τη δεύτερη συζήτηση που οργανώθηκε χθες όσον αφορά το κείμενο αυτό. Προσωπικά βρίσκω ότι είναι ένα καλό συμβαστικό κείμενο. Κατανοώ βεβαίως τον φόβο που ε, συνδέεται με μια ενδεχόμενη συζήτηση αυτού του είδους, αλλά δεν ε, συμμερίζομαι το φόβο αυτό. Όσον αφορά τα αναφερόμενα στην χάρτα, ε, δεν θεωρώ ότι το κείμενο ε, οθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μία έκκληση αντιθέτως προς την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα. Και ειλικρινά δεν κατανοώ πως στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκλογών αυτή η αναφορά στην ουδετερότητα θα έκανε οποιοδήποτε κακό. Δεν ε, θεωρώ ότι η ουδετερότητα μπορεί να είναι κακή. Και οπωσδήποτε εδώ δεν υποχρεώνουμε κανέναν για τίποτα. Επίσης, η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων δεν εκφράστηκε από αυτού. Είχαμε και συζητήσεις με τον Γκράχαμ Βότσον ως σκιώδες εισηγητές και νομίζω ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ε, αλλάζοντας δε τον ε, τίτλο κατά την έννοια που ανέφερε προηγουμένως ο Γκράχαμ, νομίζω ότι το κείμενο γίνεται ακόμα καλύτερο. Τελειώνω λέγοντας ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να ε, λέμε υψηλόφωνα τις απόψεις μας όσον αφορά την ελευθεροτυπία, την ελευθερία των μέσων στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου. Τώρα το ποιος ε, θα προσπαθήσει να ε, χειραγωγήσει τις αναφορές, μα δεν θα υπάρξει τέτοια χειραγώγηση. Εμείς έχουμε την ευρωπαϊκή αναφορά, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αναφορά αυτή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και νομίζω ότι τέτοιου είδους κείμενα με κανένα τρόπο δεν δυναμητίζουν την εκλογική διαδικασία. Το κείμενο αυτό δεν είναι ένα κείμενο το οποίο ε, έτσι χώρισε τις ομάδες, αντιθέτως τις ένωσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου μια προσωπική παρατήρηση. Εγώ θα καταψηφίσω αυτή την έκθεση, αν τελικά ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση. Εγώ ίδιος ε, είμαι εκπαιδευμένος ε, δημοσιογράφος και αν κάποιος ε, μου λέει ότι πρέπει όλοι να είμαστε ουδέτεροι, αυτό με εκνευρίζει. Όχι ουδέτεροι πρέπει να δημοσιογράφει, αλλά ανεξάρτητοι. Αυτό είναι το καθοριστικό στοιχείο. Κανείς δεν είναι ουδέτερος. Όλοι έχουν την δική τους προσωπική άποψη και σε δημόσια συζητήσεις οι δημοσιογράφοι καλούνται να αντιπαρατίθενται. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το ουδέτερο δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι ακριβώς ο αντίποδας μιας λογικής ελεύθερης κοινωνίας. Και επίσης δεν θα ήθελα αυτό που αναφέρεται στο 1α που λέει να γίνει κατανοητή η χρήση των μέσων ενημέρωση ως ε, ένα μέσο για την διάδοση των αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι το καθήκον, δεν είναι η αποστολή των μέσων ενημέρωσης ε, το ε, να είναι αντικειμενική γιατί αυτό ε, αφήνει την εντύπωση ότι καλούνται να πουλήσουν σε εισαγωγικά την πολιτική μας. Εντάξει, μπορεί να μην είναι αυτή η πρόθεσή μας, αλλά έτσι εκλαμβάνεται. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ θα καταψηφίσω και λέει να καθοριστεί επίσης ένα νομικό πλαίσιο ε, για τα μέσα ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αυτό αντίκειται στη συνθήκη, η οποία λέει ότι τα μέσα ενημέρωση εμπίπτουν σε αρμοδιότητε εθνική πολιτική. Και σε πάρα πολλέ χώρε θα έχουμε μια ε, έντονη συζήτηση για το κατά πόσο αυτά είναι η δική μα αρμοδιότητα ή όχι. Ε, δεν μπορούμε να προβάλλουμε τέτοιου είδου ε, γενικεύσει, γιατί αυτό θα ερμηνευτεί ω το ότι το Κοινοβούλιο παρεμβαίνει σε διαμάχη αρμοδιοτήτων. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά προτείνω να στηρίξουμε την κυρία Πακ ε, να στηρίξουμε λοιπόν την κυρία Πάκ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Να μην ψηφίσουμε σήμερα για αυτή την άκτηση. Αν φτάναμε στο να ψηφίσουμε, εγώ όπως σας είπα θα καταψήφιζα, αλλά Sir Graham θα προτιμούσα ε, λόγω όλων αυτών των ε, εξελίξεων να δούμε λιγάκι την όλη να βρούμε μια διατύπωση που θα μας επιτρέψει να περάσει η έκθεση. Και Sir Graham, αν θέλετε εγώ θα το κάνω αλλιώς. Ψηφίζουμε για την πρόταση της κυρίας Πάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία, από την κυρία Πακ εάν κάτι δεν έγινε σαφέ, Πριν από δύο μήνε, μου είχατε πει κυρία Πρόεδρε ότι πρέπει να μιλήσω με την κυρία Πακ για, το, για την έκθεση αυτή. Το έπραξα πριν από τρει εβδομάδε. Ε, συνέχισα τις συζητήσεις με του σκιώδει και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη αν λόγω κάποια ε, παρεξήγηση κάτι δεν πήγε πάρα πολύ καλά στι συζητήσει. Αλλά ε, εμεί προχωρήσαμε τη δουλειά μα με του σκιώδει. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ενωσιακό εργαλείο προπαγάνδας. Εδώ γίνεται λόγος ε, για ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Τώρα, εάν το πρόβλημα σχετίζεται με την ε, χάρτα των μέσων ενημέρωσης, ενδεχομένως μπορεί να κατατεθούν κάποιες τροπολογίες κατά αυτή την έννοια. Πρόεδρε, αν θέλετε, μπορούμε να καθυστερήσουμε και να το συζητήσουμε μέχρι την επόμενη φορά. Ε, και μπορούμε, προλαβαίνουμε ακόμα να το δούμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο, γιατί ε, έγινε η συζήτηση, άλλωστε πρόκειται για μια σύσταση, δεν είναι έτσι ύψης της σημασίας ε, πρωτοβουλία και νομίζω ότι καλό θα ήταν αυτό να ε, έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή η συζήτηση του θέματος να έχει ολοκληρωθεί με το τέλος της ε, ε, τωρινής θητείας. Τώρα, εάν θέλετε να το καθυστερήσουμε και αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, ας το καθυστερήσουμε. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ οι εισηγητές. Ακούσαμε προσεκτικά ε, αυτά που είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε και η κυρία Πακ και ο Σερ Γκράχαμ ε, και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια αναβολή της ψηφοφορίας ε, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Τι να κάνουμε, να το αφήσουμε για τις επόμενες μέρες. Ωραία, να το αφήσουμε γιατί ίσως είναι και δικό μου το λάθος. Ε, δεν ε, ε, είδα πολύ καλά την, την κατάσταση, δεν διάβασα πολύ προσεκτικά. Ωραία. Σας ευχαριστώ και προχωρούμε. Wir kommen jetzt zum Bericht Pakistan. Πάμε στην έκθεση Πακιστάν. Ο συνάδελφο Τσάλα είναι ο εισηγητή. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Αν όχι πάμε ευθύ αμέσω στην ε, ψηφοφορία. Er Έχω... Κύριε Στυρ. Λοιπόν πάμε στην 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 ε, το πρώτο κομμάτι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο κομμάτι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 32 σε δύο τμήματα, υπέρ, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση, ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία 16-31 το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. 33 μάλιστα. Ε, α, με συγχωρείτε, η 33 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 2 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 52 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 27, 28 εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 58 σε δύο τμήματα υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 9 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται, η 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 7 υπέρ,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 Δεβε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Δεβε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Δεβε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Δεβε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο, παρακαλώ ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γιαννάκου. Κυρία Εισηγήτρια, θέλετε να μιλήσετε, να πείτε κάτι. Από ό,τι βλέπω όχι. Περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση 36. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην ε, τροπολογία 39. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον εγκρίνεται. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 68 υπέρ, κατά Νομίζω, λέει ο πρόεδρος, ότι εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Λοιπόν, ε, αποτέλεσμα 23-23 απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 76 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η τροπολογία απορρίφθηκε με 21 προς 27. 77 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. 22 με 26 απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά νομίζω πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. «22 με 22 απορρίπτεται» ο ένας που δεν έχει την κάρτα του είναι εκείνος που τελικά από ό,τι βλέπουμε στο αποτέλεσμα της φορίας καθορίζει το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει διαφανής ε, ψηφοφορία, λέει χαριτολογώντας ο πρόεδρος. 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 83 υπέρ, κατά αποχές συμβιβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 85 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε, η 87 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 88 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η τροπολογία 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, η 93 υπέρ, κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Η ψηφοφορία έκλεισε. Προφανώς ξεκάθαρα απορρίφθηκε. Η 94 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 98 παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 22-26 απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 107 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. 18-29 απορρίπτεται. Η 108-109 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 110 υπέρ, κατά, αποχές, μισό λεπτό, η 110 παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. 22-23 το αποτέλεσμα. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 120 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Εγκρίνεται 28 με 20 το αποτέλεσμα. Συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 127 παρακαλώ. Σωστά τα λέω λέει ο πρόεδρος. Μισό λεπτό. Λάθος μου έχετε δώσει τον κατάλογο. Λάθος. Ψηφίζουμε πρώτα για την συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 134 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 142 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 38, όχι λέει ο πρόεδρος, κάνω λάθος. Πάμε στην 143, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 144, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 145 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 146 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 148 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά ε, για την 149 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση ...22 με 26 απορρίπτεται. ε, υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται ή 152 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται ή 153 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές ε, γκρίνεται. Η 12 υπέρ, κατά αποχές ε, γκρίνεται. Η 13 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 14 υπέρ, κατά αποχές ξαναψηφίζουμε για τη 13. 13, λέει ο πρόεδρος. Λάθος κάνει ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε κανένα λάθος. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. 26-22 εγκρίθηκε. Αυτή τώρα ήταν η τροπολογία 18 λέει ο πρόεδρος. Τώρα ψηφίζουμε για 18. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην Επιτροπή Πολιτισμού, παράγραφος 1. Με συγχωρείτε λέει η 3 υπέρ για την 3 κατά αποχές εγκρίνεται. Εδάφιο 1, α μάλλον, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδάφιο β, υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η Abstimmung Έκλεισε η ψηφοφορία. Der Bericht ist abgelehnt. Απορρίφθηκε η έκθεση. 21-26-1 το αποτέλεσμα. Ja. Ja. 21 Stimmen. 21 ψήφισαν υπέρ μαζί με τον κύριο Στυρ. 26 κατά. Κυρία Γιαννάκου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, με εντυπωσιάζει το αποτέλεσμα διότι στη συνάντηση που είχαμε με τους χιώδεις συγητές όχι μόνο συμφωνήσαμε στις ε, compromise ε, αλλά και στις, ε, ε, στην ειδικότερη συζήτηση δεν υπήρξαν αντιρρήσεις και θα ήθελα να γνωρίζω γιατί έγινε αυτό. Γιατί το βρίσκω ανακόλουθο σε σχέση με τη συνεννόηση που είχαμε κάνει. Κυρία Γιαννάκου, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ίσως οι σκιώδες ηγητές δεν έπισαν τις πολιτικές τους ομάδες. Εγώ το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να επικυρώσω είναι το αποτέλεσμα. Νικολάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων στην τελευταία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών ζητήσαμε την κυρία Γιαννάκου να αποσύρει την προφορική τροπολογία 16 και είπαμε ότι αν περάσει αυτή η τροπολογία συμβιβασμού θα καταψηφίσουμε το σύνολο. Χθε στον κατάλογο ψηφοφορίας βάλαμε μια κόκκινη γραμμή για την συμβαστική τροπολογία 16. Αυτό ήταν απόλυτα σωστό και δίκαιο. Είπαν, είπαμε ότι αυτή ήταν η άποψη της ομάδα μα και το κάναμε σαφέ. Τάνοκ. Εμεί δεν είχαμε πρόβλημα με τη 16, είχαμε πρόβλημα με τις τροπολογίες για την ενιαία έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πέρασαν. Αυτό ήταν κομβική, ε, τροπολογίες για μας. Γι' αυτό εμείς κρατήσαμε στάση αποχής. Θέματα όπως η έδρα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αυτό επίσης δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, δυστυχώς. Μα αυτό είναι διαφορετικό το η ενιαία έδρα με τα πολιτιστικά θέματα, λέει ο πρόεδρος. Πώς σχετίζεται το θέμα αυτό με την έκθεση αυτή. Τι έχει η ενιαία έδρα με την ε, πολιτιστική διπλωματία. Είναι η πολιτιστική κατάσταση της Αλσατίας ίσως που σας ενδιαφέρει. Α, έχει να κάνει με κάποιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει ο πρόεδρος. Συμβουλή Ασφαλείας του λέει γραμματεία. Κατανοώ. Νομίζω ότι είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεπλέκεται. Νομίζω κύριε Τάνοκ ότι ήταν το θέμα της ενίας της μοναδικής έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οδήγησε σε όλα αυτά. Πάση περιπτώσει αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λόγω δύο θεμάτων Το ένα ήταν το θέμα της ενιαίας έδρας ή της παρεξής γύρω από την ενιαία έδρα ε, και το άλλο ήταν η συμβαστική τροπολογία 16. Μπορούμε να επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα και να ξαναδοκιμάσουμε έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Ερχόμαστε τώρα στην αντιπυραυλική ασπίδα. Ο κύριος Τέρχο θέλει να πει κάτι. <clears throat> Όχι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Χρειάστηκε πολύ εργασία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην ε, τελική μορφή αυτής της έκθεσης. Αλλά στο τέλος καταφέραμε να έχουμε μια ευρεία συνένωση για το θέμα αυτό Το αρχικό κείμενο πιστεύω ότι θα ήταν πιο απλό, αλλά επειδή ήταν δύσκολα τα πράγματα και μέσα στο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν δύσκολο να επιλύσουμε όλα τα θέματα αυτά. Και επειδή δεν θέλαμε να χάσουμε την ευκαιρία αυτής της έκθεσης, καταλήξαμε σε μια συνένεση, σε μια συμβαστική θέση για την έκθεση αυτή που βασίζεται σε μια σειρά ε, Συμβαστικό τροπολογιό και φυσικά και η Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας έχει συμφωνήσει για όλα αυτά. Ωραία, ξεκινάμε την ψηφοφορία. <clears throat> Συμβιβαστική τροπολογία 5, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην παράγραφο υπαριθμό 3 <clears throat> του αρχικού κειμένου. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σύμβαστη 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Σύμβαστη 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 6 του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 51 και 52 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 53 εκπίπτει συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68, 69 και 70 είναι, είναι ταυτόσιμες των τριών εισηγητών. Ψήφι υπέρ. από τον κύριο Λίζεκ και όχι από τον κύριο Πάσκου. Για τον κύριο Λίζεκ και όχι τον κύριο Πάσκου αυτό που έκανε το σχόλιο. Γίνεται δεκτή τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 και 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 89 και 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ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 τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 38 ψήφι υπέρ, 8 κατά με 3 αποχές. Γίνεται δεκτή. Εντάξει, συγχαίρουμε τον συγητή. έχουμε τελειώσει τις ψηφοφορίες. Κύριε Σούλτς. κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου θα συντάξει μια έκθεση μειοψηφία για το θέμα αυτό. Κυρία Λέζινγκ, και για τη δική μου πολιτική ομάδα θα συντάξουμε μια έκθεση μειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαίρω τον εισηγητή όπως είπα προηγουμένως. Σημείο 18 τώρα. Η έκθεση για την Τουρκία. Έκθεση πρόοδου για την Τουρκία. Ζήτω από την κυρία Ρία Όμεν να λάβει το λόγο. Yep. Yeah. Uh, chairman. Κύριε Πρόεδρε, ε, πολύ πηγενέλα έχει η αίθουσα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ήδη την 9η Δεκεμβρίου είχαμε μία πρώτη συζήτηση για το σχέδιο ψηφίσματος για την Τουρκία στην Επιτροπή μας. Λίγο θα ήταν να πούμε ότι υπήρξαν κάποιες εξελίξεις εντωμεταξύ. Ως εισηγήτρια για την Τουρκία ποτέ δεν ησυχάζω και ποτέ δεν βαριέμαι. Λέω λοιπόν ότι μας απασχολούν ιδιαίτερα οι πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε την τελική μορφή του ψηφίσματος έτσι ώστε και να σκεφτούμε περισσότερο και να αντικατοπτρίζει το κείμενο την πραγματική κατάσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντιμετώπιση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του κράτους δικαίου και της λειτουργίας του. Περιμένουμε λοιπόν, προσδοκούμε ότι οι διαδικασίες που ξεκίνησαν την 7η Ιανουαρίου θα συνεχίσουν. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις μας έχουν προκαλέσει προβληματισμό όσον αφορά την ε, ακαιρεότητα και την ε, αμεροληψία όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές. Όσον αφορά τώρα την, ε, τους κανόνες που διέπουν το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων, πρέπει να πω ότι μας απασχολεί επίσης οποιαδήποτε κίνηση ε, αύξησης του ρόλου και της, του Υπουργείου Δικαιοσύνης ε, μας απασχολεί ακόμα περισσότερο. Επομένως, ζητούμε από την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει οποιαδήποτε παρέμβαση στις δικαστικές διαδικασίες και να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της, ε, του διαχωρισμού των εξουσιών, καθώς ε, και ότι ε, γίνονται σεβαστά τα σχετικά άρθρα του συντάγματος. Καλούμε δε τις ε, τουρκικές αρχές ιδιαιτέρως να λάβουν υπόψη την, τους κανόνες της Επιτροπής της Βενετίας. Κύριε Πρόεδρε, το, η πρόταση ψηφίσματος εξέφραζε τους προβληματισμούς όσον αφορά την ελευθεροτυπία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία. Οι πρόσφατες εξελίξεις, ας πούμε η, έγκριση του νόμου για το ίντερνετ την προηγούμενη εβδομάδα, ε, καθώς επίσης και η απόλυση ε, δημοσιογράφων, καθώς επίσης ε, και η, αρχή διαδικασιών κατά ξένων δημοσιογράφων, ε, δυστυχώς επιβεβαίωσαν τους προβληματισμού μα. Ως Ευρωπαϊκό επανειλημμένα ε, έχουμε ζητήσει από την ε, Τουρκία ε, να τροποποιήσει τον νόμο 5651 του 2007 όσον αφορά το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Ε, διότι είναι ένας νόμος ο οποίος περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, ε, μειώνει το δικαίωμα πρόσβασης στο ίντερνετ, το δικαίωμα των πολιτών, ε, καθώς επίσης έχει δυσανάλογο πεδίο εφαρμογής. Επίσης θεωρούμε ότι τέτοιου είδους κινήσεις αποτελούν, αποτελούν παράβαση της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, αντιθέτως, είδαμε ε, κάποιες τελευταίες κινήσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν απαλύνουν τους προβληματισμούς μας, αντιθέτως τους εντείνουν επί περαιτέρω. Κύριε Πρόεδρε, Όντω την, πρώτη εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση μεταξύ, μεταξύ σκιωδών εισηγητών. Αυτή έλαβε χώρα στο Στρασβούργο και είμαι απολύτως πεπισμένη ότι μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο έκφρασης των προβληματισμών μας όσον αφορά το θέμα αυτό. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης καθώς επίσης ε, και τον ε, υπεύθυνο των πολιτικών για την οικογένεια Σαμπταλά Χεργίν. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά τα θέματα που μας απασχολούν. Επίσης, καλωσορίζω του, τις προσπάθειες του Καβούσογλου όσον αφορά την προσέγγιση της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πρέπει να σας πω ότι θέλω να τελειώσω τη σημερινή μου παρέμβαση με κάτι θετικό. Χαίρομαι γιατί οι διαδικασίες, οι διαπραγματεύσεις για την Κύπρο ξαναξεκίνησαν και ευελπιστώ ότι θα οδηγήσουν σε μία διαρκή λύση θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην χρησιμοποιήσουν το ψήφισμα για την Τουρκία σαν ε, πλατφόρμα ε, μέσω της οποίας ε, θα εμπλακούν ακόμα περισσότερο και θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο οι διαδικασίες. Ζητούμε οπωσδήποτε εντόνως ε, την ε, λύση, ε, τη συνένωση, της, την επανένωση μάλλον της Κύπρου. Ζητούμε μια βιώσιμη λύση βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία σας. Ο κύριος Σομπιόλς, αυτή η έκθεση αντιμετωπίζει μια χρονική περίοδο η οποία σημαδεύτηκε από μια σειρά κινητοποιήσεων, από συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, σκάνδαλα στη δημόσια ζωή της Τουρκίας. Για τους λόγους αυτούς η δική μας πολιτική ομάδα πιστεύει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις βασικές αρχές που διέπουν πάντα τη στάση μας. Καταρχήν, στεναρότητα σε ό,τι αφορά την προάσπιση των στόχων μας και των απαιτήσεών μας, τόσο σε ό,τι αφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Τουρκίας για τις ε, μεταξύ των δύο πλευρών σχέσεων. Δεύτερον, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα αντικειμενικό και επακριβή χαρακτήρα στις αξιολογήσεις σε σχέση με την κατάσταση της δημόσιας ζωής στην Τουρκία και τρίτον θέλουμε να εστιάσουμε ιδιαίτερα για να μπορούμε να αντλήσουμε τα σωστά συμπεράσματα, να μπορέσουμε να προσέξουμε τα μηνύματα τα οποία πρέπει να απευθύνουμε και στα κράτη-μέλη της Ευρώπης και στην ίδια την Τουρκία σε σχέση με το πάρα πολύ δύσκολο θέμα του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την υποστήριξή μας στη γενική μας γραμμή που είναι η υποστήριξη των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία προς την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του τύπου, γενικά δηλαδή την υποστήριξη που έχουμε προς τον δημοκρατικό πλουραλισμό στην Τουρκία. Έχουμε μια θετική αξιολόγηση για το σχέδιο έκθεσης και για τις συμβαστικές ε, τροπολογίες και λύσεις που έχουμε επιτύχει. Δεν έχω καμία αμφιβολία, θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε μια ευρεία πλειοψηφία γύρω από αυτή την έκθεση όταν ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, λέει Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, Λέω, κύριος ε, Λάμστροφ, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγητρία συγγνώμη, για την πάρα πολύ επαγγελματική και ικανή εργασία της στο Στρασβούργο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ιδιαίτερα καρποφόρα συζήτηση για διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν επεξεργασία, διότι υπήρχαν διαφορετικέ απόψει μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά έχουμε βρει ένα σωστό πιστεύω δρόμο. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά, όπου έχουμε μια γενική συνένεση, απλώς θα σταθώ σε ορισμένα σημεία όπου θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε περισσότερο την ε, έκθεση αυτή. Καταρχήν, η δική μας άποψη είναι ότι τα γεγονότα του τέλους του έτους ε, δεν συνάδουν με την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπενχάγης στη χώρα αυτή υπήρξαν όλες αυτές οι υποστηρίζουν να τονίσουμε τα κριτήρια της Κοπεχάγης ότι με τις διαμαρτυρίες αυτές και τις διαδηλώσεις γίνεται πιο σαφές ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ελευθερία σε, για τους δικηγόρους, για τους ε, ιατρούς, που υπάρχει κίνδυνος να περιοριστούν οι δυνατότητές τους και αυτό αναφέρεται και σε άλλα σημεία στην έκθεση. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο νομίζω πρέπει να αντιμετωπιστεί και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ίσως λιγάκι πρωτού εξετάσουμε αυτό το θέμα πριν από την ψηφοφορία την τελική. Πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε ρεαλιστές και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο τάσεων στην Τουρκία. Από τη μία μεριά το συντηρητικό ΑΚΠ, το κόμμα της εξουσίας, και από την άλλη μεριά η λεγόμενη κίνηση Χισμέτ, η κίνηση της υπηρεσίας, όπως λέγεται, του Φέτουλα Γιουλέν. Και νομίζω ότι το κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια έκκληση προς την κίνηση Χισμέτ να εξασφαλίσει την διαφάνειά της και επομένως το κίνημα αυτό το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον Φέτιουλαχ Γιουλέν και εμπνέεται από αυτόν, οι εκπρόσωποι του κειμένου ε, του, της, της κινήσεως αυτής να μπορέσουν να είναι έτοιμοι να εξηγήσουν σε τι συνίσταται το κίνημα Χισμέτ, ποιοι είναι οι στόχοι του, διότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα με το οποίο έχουμε ήδη ε, καταπιαστεί ως ε, Επιτροπή. Υπενθυμίζω την ε, σύλληψη του Αχμέτ Σίκ και του κυρίου Σενέρ, του συναδέλφου του, όπου έγινε σαφές ότι υπήρχε μια πίεση από το κίνημα Χισμέτ στην αστυνομία και στην ε, δικαιοσύνη και επομένως το κίνημα αυτό έχει κάποιο ρόλο μέσα στην ε, κρατική μηχανή της Τουρκίας. Καλέσαμε τον Αχμέτ για να μας παρουσιάσει τις απόψεις για τα θέματα αυτά. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη ε, συνάντηση. Εάν λοιπόν είναι το κίνημα Χισμέτ έτοιμο να δώσει περισσότερες εξηγήσει και μεγαλύτερη σαφήνεια, εγώ δεν βλέπω γιατί το κοινοβούλιο μας δεν θα πρέπει να περιλάβει μια τέτοια έκκληση στην εκθεσή του, ώστε να γίνει μια τέτοια διευκρίνηση και λυπάμαι που η συγγήτρια μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί αυτή την ε, αίτησή μας. Ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό για μας ως φιλελεύθερους είναι το θέμα του πλουραλισμού. Η δημοκρατία δεν είναι μονάχα οι εκλογές. Μια πλειοψηφία δεν έχει αυτόματα και το δικαίωμα να ε, ξεχνάει τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να προσπαθεί να ομοιογενοποιήσει όλες τις μειονότητες. Η διασταυρούμενη έλεγχη σε μια δημοκρατία είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται μονάχα στην εκλογική διαδικασία. Και ένα τελευταίο σημείο ο νόμος για την ε, λογοκρισία ουσιαστικά στο ίντερνετ, ο οποίος έχει μόλις εγκριθεί αμέσως μετά την ε, επίσκεψη του κυρίου Ερντοάν στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, είναι ένας νόμος ο οποίος είναι σε μετοπική αντιπαράθεση με τις αιτήσει των υπερμάχων της ελευθερίας έκφρασης. Είναι και μία ακόμα εξέλιξη η οποία πρέπει να αντανακλάται κατά τη δική μου άποψη σε, στην έκθεση αυτή και συμφωνώ με τη Ρία σε αυτό ότι χρειαζόμαστε και λίγο χρόνο για το θέμα αυτό. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω να έρχεται ο Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο να λέει τα πράγματα πάνε μια χαρά και αυτό το οποίο συμβαίνει παράλληλα είναι το τουρκικό κοινοβούλιο να εγκρίνει ένα τέτοιο νόμο για το ίντερνετ το οποίο αντιβαίνει προ τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πολύ στην Τουρκία είπαν ότι αυτός ο νόμος ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα. Μα είναι ένας νόμος, λέει ο κύριος Λάμστορφ, που μπορεί να έχει κάποια στοιχεία από ευρωπαϊκές νομοθεσίες, αλλά τελικά καταλήγει στο να είναι μία ε, μορφή λογοκρισίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Ερντοάν. Εντάξει, αυτό δεν αναπόκειται, σε, σε να ε, να κρίνουμε. Ο κύριος δεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι... Ε, με όλες τις αντιπροσωπείες και τα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβούλιο είναι σαφές ότι υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις για την Τουρκία και υπάρχουν θέματα τα οποία είναι σημαντικά ε, για διάφορα μέλη, διαφορετικά θέματα για τον καθένα αυτό το ομολογώ και Καταλαβαίνω την άποψη συναδέλφων, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν αναφερόμαστε στο ε, θέμα της Κύπρου και δεν το περιγράφουμε σωστά. Η ιστορία στρεβλώνεται συστηματικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση. Και γνωρίζουμε πολύ καλά το λόγο γιατί. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν και άλλοι τομείς ε, διστάμενων ε, απόψεων. Κατανοώ ότι υπάρχουν, όπως σας είπα, διαφορετικές απόψεις. Αν δούμε λιγάκι το τι συνέβη κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν τραγικά γεγονότα, ε, τρινήσαμε πολλά θύματα και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ατυχές το γεγονός το να συνεχίζουμε να χαρακτηρίζουμε αυτά τα γεγονότα ως γενοκτονία, το οποίο όπως ξέρετε πολύ καλά έχει μια πολύ συγκεκριμένη νομική ερμηνεία στα Ηνωμένα Έθνη και αυτό προφανώς αφορά την σκόπιμη, ε, τον εξαντραποδισμό, την εξαφάνιση ε, συγκεκριμένου λαού. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό ισχύει και το να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια αυτό είναι ιδιαίτερα προσβλητικό για τους ε, Τούρκους ε, συναδέλφους. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ που έχει παρισφρήσει στην έκθεση αυτή η ορολογία. Ε, κοιτάξτε, έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες, κατανοώ τις προσπάθειες της ΡΙΑ να καταλήξει σε συμβασμού, σε κάποιους τομείς το κατάφερε αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι δεν είναι κακή έκθεση, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία χρήζουν βελτιώσεων. Ε, η κυρία εισηγητής ε, μας έχει φέρει μια ισορροπημένη έκθεση όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Σε γενικέ γραμμέ θεωρώ ότι η προσπάθεια που έγινε ως προς τις συμβαστικές τροπολογίες είναι ικανοποιητική. Ε, δεν θα αναφέρω πολλά, ε, συντάσσομαι με τις απόψεις του συναδέλφου κ. Λάμπστορφ ε, και θεωρώ ότι οι αναφορές στην αναγκαιότητα ύπαρξη ανεξάρτητου δικαστικού κλάδου και διάκριση των αξιών είναι απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξη ενός κράτους δικαίου που πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Ε, τα όσα προσφάτως έγιναν στην Τουρκία πρέπει να μας προβληματίσουν και να μας ε, δημιουργήσουν ερωτηματικά κατά πόσον η παρεμπόδιση από την κυβέρνηση της ελευθερίας του τύπου και της εκπροσώπης άλλων πολιτικών δυνάμεων δείχνουν ότι η πορεία της Τουρκίας προς μια δημοκρατία δυτικού τύπου είναι ακόμη μακρά και απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ως προς τις συμβαστικές αναφορές που αφορούν το άνοιγμα κεφαλαίων θεωρώ ότι από τη στιγμή που η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιαδήποτε συζήτηση για την ευρωπαϊκή τη προοπτική δεν έχει πρακτικό νόημα. Είναι απαραίτητο η Άγκυρα να αντιληφθεί και να παραδειχθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα 28 ισότιμα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ω προ το άνοιγμα του κεφαλαίου 15 για την ενέργεια. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΕΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, ενώ παράλληλα δεν αναγνωρίζει και ούτε σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών για την έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων. Ω εκ τούτου δεν νομίζω ότι είναι φρόνιμο το άνοιγμα του κεφαλαίου υπό τι παρούσε συνθήκε. Πρέπει να αντιληφθούμε και το φοβάμαι αυτό ότι το εσωτερικό πρόβλημα της Τουρκίας που αυτή την εποχή ογκούται ε, πρέπει να περιοριστεί στα όρια αυτής της χώρας και πρέπει να συνδράμουμε να περιοριστεί και να μην εξαχθεί στο εξωτερικό με επιθετικές ενέργειες κατά γειτόνων και μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ω προ το πνεύμα τη συμβαστική τροπολογία 12 για τη θρησκευτική ελευθερία είναι και η τροπολογία μου υπαριθμών 200 που αναφέρεται στι δηλώσει και ενέργειε Τούρκων αξιωματούχων για μετατροπή του ναού τη Αγία Σοφία σε τζαμί που αποτελεί παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι η συζήτηση φέτος για την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας στο Κοινοβούλιο συμπίπτει σήμερα με την έναρξη νέας διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού στη Λευκοσία. Θεωρώ σημαντικό να σας πω και να γνωρίζετε ότι το κόμμα μου, το ΑΚΕΛ, ε, που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, στηρίζει ε, τις προσπάθειες της, ε, που καταβάλλονται σήμερα για επίλυση του Κυπριακού. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι στηρίζεται, επαναλαμβάνω, αυτή η διαδικασία από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά τις όποιες επιφυλάξεις έχουμε για το κοινό ανακοινωθέν. Ε, προς αυτήν την κατεύθυνση καλούμε όλους όσοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του Κυπριακού να το κάνουν. Θεωρώ δε σημαντικό το ότι για πολλωστή φορά η ραπορτέρ ε, αναζητά την παράδοση της πόλης της Αμοχώστου <clears throat> στην Κυπριακή Δημοκρατία που την κατέχει η ε, ο τουρκικός στρατός. Ε, εάν αποδοθεί η πόλη της Αμοχώστου ή αποδιδόμενη η πόλη της Αμοχώστου στους κατοίκους της, όπως το ζητά η κυρία Ούμεν και το Κοινοβούλιο για τόσα πολλά χρόνια, θα δώσει μια τεράστια όθηση ε, προς την κατεύθυνση της επίλυσης. Και όσοι ενδιαφέρονται για την επίλυση πρέπει να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η έκθεση για μας έχει θετικά και αρνητικά και θα τα αναλύσουμε ε, ολοκληρωμένα στο τέλος για να δούμε την στάση που θα τηρήσουμε. Ε, θεωρούμε σημαντικό επίσης να πούμε ότι στις συμβιβαστικές τροπολογίες δυστυχώς δεν υπάρχει αναφορά α, φέτος στον επικισμό και καλούμε την, ε, η συγγήτρια να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Κλείνω λέγοντας ότι τα κεφάλαια 23-24 που ζητά η ραπορτέρ να ανοίξουν δεν μπορεί να ανοίξουν εφόσον η Τουρκία δεν υλοποιεί συγκεκριμένες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με, το, με τα συγκεκριμένα κεφάλαια. Ευχαριστώ και καλώ ξανά όλους, επειδή ξεκινά σήμερα μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, να είναι ιδιαίτερα επικοδομητική υπέρ αυτής της προσπάθειας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Όμεν Γόιτεν, διότι περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια τα προβλήματα. Εμείς ε, έχουμε προσδοκίες εναντί της Τουρκίας και πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένη συμφωνώ με την έκθεση και με τον τρόπο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση στην Τουρκία. Έχω κάποιες ανησυχίες, όπως και η συγγήτρια, διότι στην έκθεση γίνεται λόγος για ε, προβλήματα στα Βαλκάνια που δεν έχουν επιληθεί, για προβλήματα που υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στην Τουρκία και τη Βουλγαρία και εμείς αυτό το έχουμε αναφέρει επανειλημμένα σε διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά δεν έχουν υπάρξει αντιδράσεις εκ μέρους της ε, τουρκικής κυβέρνησης η οποία η τουρκική κυβέρνηση ναι, λέει ναι βέβαια θέλουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα αλλά δεν κάνει τίποτα και έχουμε αποκομίσει την εντύπωση ότι οι Τούρκοι πολιτικοί ε, θέλουν να επαναπροσδιορίσουν τα σύνορα στα Βαλκάνια. Γιατί υπάρχουν ε, τέτοιες ε, απόψεις. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να επανέλθουν τα σύνορα όπως ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε δημιουργεί ένταση στα Βαλκάνια, δημιουργεί προβλήματα και είναι σαφές ότι για το λόγο αυτό τίθενται επιτάπητος και άλλα θέματα, ας πούμε, η ανεξαρτησία των λαών της, των Βαλκανίων. Τι θα γίνει με την ανεξαρτησία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια ε, ακολουθεί μια πολιτική διεύρυνσης, αλλά θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Το τουρκικό κράτος έχει διαφορετική άποψη Όσον αφορά τις ε, αδειοδοτήσεις, τη χορήγηση, μάλλον ε, τη δυνατότητα διέλευσης ε, φορτηγών μέσω του τουρκικού εδάφους. Απαγορεύεται πλέον αυτό. Τα δικά μας τα βουλγαρικά φορτηγά δεν μπορούν πλέον να διέλθουν από τουρκικό έδαφος. Προφανώς και θέλουμε να στηρίξουμε τις συμβαστικές προτάσεις, αλλά πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για το λόγο αυτό, εγώ έχω καταθέσει τροπολογίες και παρακαλώ πολύ να τις λάβετε υπόψη, γιατί νομίζω ότι οι δικές μου οι τροπολογίες είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούτε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρία Όμεν για την ρητή και ξεκάθαρη αναφορά της στην αναγκαιότητα επίλυσης του κυπριακού προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Γιατί μόνο έτσι η λύση θα είναι βιώσιμη. Αν δεν είναι δίκαιη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη κυρία Όμεν. Υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος στην τροπολογία 259, την οποία έχω καταθέσει με μια άλλη συνάδελφο, η οποία νομίζω είναι, αρκετά σημαντικό, είναι καθαρά ε, τυπογραφικό το λάθος και θα παρακαλούσα πολύ να διορθωθεί και να ληφθεί υπόψη στην διόρθωση. Όπως σας έχω πει είναι το Amendment 259 και λέω calls on Turkey to immediately... Ζητά από την Τουρκία να αποσύρει άμεσα τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να μεταφέρει την πόλη της Αμοχώστου στους νόμιμους κατόχους της. Την περίκλειστη περιοχή της ε, Αμοχώστου, την ε, πόλη της Αμοχώστου σε αυτή την περίπτωση. Επιστρέψει την πόλη της Αμοχώστου στους νομίμους κατοικούς της ως ένα ελάχιστο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης Θεωρώ ως πολύ σημαντική τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προσπάθειες για βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος και ιδιαίτερα την ρητή αναφορά στο ότι η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αποκλήσεις από το κοινοτικό κεκτημένο. Ωστόσο, παρόλο που αυτή τη στιγμή ξεκινούν οι συνομιλίες στη Λευκοσία, η Τουρκία έχει δώσει τη δική της ερμηνεία για το κοινό ανακοινωθέν η οποία ερμηνεία ουδεμίαν σχέση έχει με την ερμηνεία που δίνει η Κυπριακή κυβέρνηση. Έχω καθήκον να υπερασπίζομαι την Κυπριακή Δημοκρατία και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο σας θυμίζω και τις δικές σας υποχρεώσεις απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης αδύναμο και εκτεθειμένο, σε απειλές. Δεν αναφέρεται καθόλου οτιδήποτε κυρία Όμεν για τον επικισμό και τονίζω ότι το κεφάλαιο 15 δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να δεχθεί να ανοίξει με το τουρκικό ναυτικό να περιπολεί μέσα στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε τόσο προσεκτικά. Uh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ομολογήσω ότι μέχρι τώρα ή τέλος πάντων μέχρι πριν από λίγο ε, δεν είχα άποψη έτσι πολύ έντονη όσον αφορά τα θέματα της ε, Τουρκίας. Ε, τους τελευταίους μήνες ωστόσο είχαμε πολλά καινούρια στοιχεία. Θα θυμούνται οι συνάδελφοι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ή τέλος πάντων την προηγούμενη δεν θυμάμαι ήρθε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας και μας επισκέφθηκε ε, και με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο στην συνέντευξη απάντησε σε κάποια μελήματα ε, τα οποία ήταν πολλά και διάφορα και αυτό βεβαίως από μόνο το είναι ανησυχητικό επίσης ε, υπάρχουν και κάποια, κάποιοι προβληματισμοί όσον αφορά ορισμένα στοιχεία του τουρκικού συντάγματος που δεν έχουν ακόμα λυθού. Θα ήθελα πάντως και εγώ να συγχαρώ την κυρία Ούμεν Ράιτεν για τον επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί το θέμα. Αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσε μπορούσε να σχολιάσει, όχι ακριβώς να απαντήσει, επί τριών ε, σημείων που ήθελα να θίξω. Ένα, έχει πραγματικά ε, στοιχεία ή μαρτυρίες ε, σχετικά με το κατά πόσον πραγματικά θέλει η τουρκική κυβέρνηση να ε, προχωρήσει σε ένταξη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πραγματικές μαρτυρίες, πραγματικά στοιχεία. Δεύτερο, βλέπει να υπάρχουν κάποια πραγματικά στοιχεία, κυρίως και στον απόϊχο της επίσκεψης Ερντογάν, στοιχεία λέω βελτίωσης σε σχέση με την ε, ολοένα και ε, ε, επιταχύρω βένουσα κατάσταση των τελευταίων μηνών τουλάχιστον όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και τα λοιπά. Τρίτον, και ξέρω ότι αυτό απασχολεί πολλούς συναδέλφους διαρκώς, υπάρχουν οποιαδήποτε πραγματικά στοιχεία στη στάση της κυβέρνησης ε, ε, όσον αφορά την κατάσταση με την Κύπρο. Μήπω Μήπως υπάρχει έτσι μία μεταστροφή τύπου Αγίου Παύλου, ε, κάποια φώτιση ξαφνική για να αλλάξει, ε, για να αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά ή τη στάση της όσον αφορά την ε, ε, Κύπρο. Ε, δεν ξέρω εάν στην παρούσα συγκυρία πραγματικά κάνει τα πάντα για να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θέλει πραγματικά να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει μία γενική επιθυμία, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πω ότι το ΑΚΠ του Πρωθυπουργού ε, έμαθα ότι <laughs> είναι στην ίδια πολιτική ομάδα που βρίσκομαι και εγώ. Και αυτό πρέπει να σας πω ότι πολύ με προβλημάτισε. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να είμαι στην ίδια πολιτική ομάδα με το ΑΚΠ, Εκτός κι αν η κυρία Όμεν Ρόιτερ καταφέρει να με πείσει ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία μεταστροφής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια εξ ονόματο τη ε, ομάδα μου. Έκανε μια πολύ καλή δουλειά ε, μέσα σε, ε, για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, σε χαλεπούς καιρού, καιρούς κρίσης και τα λοιπά. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι και λόγω τη της των αγορών και λόγω της σύραξη στη Συρία τα προβλήματα έχουν γίνει διεθνή και έχουν γίνει πολύ πιο έντονα Βεβαίω Βεβαίως ε, θα πρέπει να ε, ε, προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία έτσι ώστε να βρεθεί η άκρη όσον αφορά αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς και να δούμε και ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος των Ισλαμιστών κτλ. Ξέρουμε ότι με το Ισραήλ οι σχέσεις ήταν καλές παλιότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, τώρα τα πράγματα έχουν ε, ε, αλλάξει. Υπάρχουν και υπόνοιες για στήριξη των αντιμαχόμενων των Ασάντ στη Συρία. Η κατάσταση με την Κύπρο είναι αυτή που είναι και δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δεν φαίνεται να προχωρούν και οι διαδικασίες όσον αφορά την εξέβρεση μιας μόνιμης μόνιμης και ειρηνικής ε, λύσης. Ε, αυτά θυμίζουν και άλλες καταστάσεις και άλλες συζητήσεις. Ε, τα πράγματα έχουν αλλάξει μετά από την αρχή εξορίξεων για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας πω ότι θα ήθελα να στην τροχιά των όσων είπε ο συνάδελφος ε, Βανόρντεν. Ε, υπάρχει η τροπολογία μου 158 ε, στην οποία αναφέρω την θέση της τουρκικής κυβέρνησης όσον αφορά την μνημόνευση της, αρμενικής, της γενοκτονίας των Αρμενίων και δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση αυτού του όρου γιατί βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και άλλωστε υπήρχε μια μια, ένας γενικευμένος διωγμός των χριστιανών, ε, αλλά Πρέπει να πω ότι η δική μου τροπολογία 158 είναι μάλλον μια αναγνώριση ε, του ε, γεγονότος ότι δεν προσπαθεί πλέον ε, η τουρκική κυβέρνηση να καταδικάζει ή να σέρνει ενώπιον των δικαστηρίων όλους αυτούς που αναφέρονται στην γενοκτονία και τους διωγμούς των χριστιανών κτλ. Επίσης θα ήθελα να αναφερθούμε και στα δικαιώματα των χριστιανών στην Ανατολική Τουρκία των Ασυροχαλδαίων στην Ανατολική Τουρκία. Ε, υπάρχουν προβλήματα και με αυτές τις ε, μειονότητες. Ε, νομίζω ότι αυτά και εμείς θα στηρίξουμε την έκθεση. Η κυρία Γιαννάκου παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως πάντοτε η κυρία ουμεν έχει εκπονήσει μια έκθεση εξαιρετικά συνεπή προς τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βέβαια ξέρω ότι πολλές φορές δεν θέλει να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα αλλά δυστυχώς στην περίπτωση της Τουρκίας δεν υπάρχει πρόοδος στα βασικά που έχουν σχέση ε, με την πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι η αποδοχή της Άγκλος, είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας και η κατοχή της Κύπρου, ε, είναι οι συνεχείς παρεμβάσεις ε, στα θέματα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών ε, και υπεράνω των, της θάλασσας του Αιγαίου και των ελληνικών νήσων, δηλαδή όλα όσα δεν πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει συνθήκες καλής γειτονίας. Πολλοί αμφισβητούν την διάθεση της Τουρκίας πλέον να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Τουρκία θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι, χωρίς να αλλάξει αυτά που συνιστούν τον βασικό πυρήνα κυριαρχίας και εξουσίας της στην περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κατανοηθεί από όλους μας. Και φυσικά η έννοια της, του ανοίγματο των κεφαλαίων <clears throat> για μένα δεν πρέπει να υπάρξει η Τουρκία εάν δεν δεχτεί να αναγνωρίσει το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να προχωρήσει τα θέματα ε, ε, του οδικού χάρτη της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κυρία Όμεν, ελπίζω ότι και οι τροπολογίες μας θα έχουν καλή τύχη από δική σας πλευράς για να ικανοποιηθούν και ορισμένα ζητήματα στα οποία υπάρχει ευαισθησία. Ευχαριστώ πολύ. Οφείλω να χαιρετήσω την προσπάθεια της εισηγήτριας και ταυτόχρονα να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τη σημερινή της τοποθέτηση, δηλαδή ότι έχουμε νέες εξελίξεις στην Τουρκία και το ζήτημα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Η δική μου άποψη είναι ότι η συγγήτρια επί της ουσίας δεν μπαίνει σε βάθος σε αρκετά ανοιχτά ζητήματα που ουσιαστικά αντιστρατεύονται τη διεθνή ενόμη Τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτημένο. Εξηγούμε. Δεν καταδικάζεται ξεκάθαρα, όχι απλά διακηρυχτικά, η εισβολή και η κατοχή μιας χώρας που είναι πλήρες μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καμιά ουσιαστική ξεκάθαρη αποδοκιμασία πως η Τουρκία συνεχίζει τον παράνομο επικισμό. Καμία ξεκάθαρη θέση για το ότι η Τουρκία δεν ανεγνώρισε την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά την προεδρία της και κατ' επέκταση την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς συνεχίζει η Τουρκία να απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αφημώνει τον τύπο όπως έχει λεχθεί την ελευθερία να φυλακίζει παράνομα δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, πνευματικούς ανθρώπους, καταστέλει βία της κινητοποιήσεις απεργών του τουρκικού λαού, διώκει τους χριστιανούς ανοιχτό το κουρδικό ζήτημα. Η έκθεση επιτέλους πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην είναι απλά μια περιγραφή ή ακόμη και διακήρυξη. Όσο χαϊδεύουμε την Τουρκία, άλλο τόσο δυναμητίζουμε και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του τουρκικού λαού. Και βέβαια τέλος, σαν ένα πρώτο βήμα πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι ότι δεν μπορεί να ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φιλορή από τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης. Καλημέρα. Η πρώτη συζήτηση για αυτή την έκθεση έγινε το Δεκέμβριο και τότε είχα την χαρά να παρουσιάσω τα σχόλια της Κομισιόν σε συγκεκριμένα θέματα που αναφέρονται στο σχέδιο της έκθεσης. Πράγματι υπήρξαν ανησυχητικέ ε, εξελίξεις όπως ελέγχθη από τότε που ήμουν ενώπιον σας το Δεκέμβριο. Υπήρξε η απάντηση της ε, τουρκικής κυβέρνησης της ε, ανακρίσεις για διαφθόρα μετά την 17η Δεκεμβρίου και όλα αυτά είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ανακριτικών αρχών και της αστυνομίας. Ο Επίτροπος Φίλου από την αρχή εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για αυτές τις εξελίξεις και τόνισε προς τον Υπουργό Εξωτερικών Νταβούτογλου και τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τσαβούσογλου ότι είναι απαραίτητο ο σεβασμός για τον νόμο και η διάκριση των εξουσιών που είναι βασικές αρχές της δημοκρατίας και κέρυες για τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας. Ο Αντίδροπος Φίλε τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε καταγγελίες για διαφθορά με αμερόληπτο και διαφανή τρόπο. Θα πρέπει αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να απόσχει δράσεων οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητα των ενεξελίξη ερευνών. Η Κομισιόν έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πλαίσιο στο σχέδιο νόμου για τη δικαστική εξουσία που όπως είπατε έχει διατάξεις οι οποίες έχουν σαν στόχο να αλλάξουν τη λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Εισαγγελών και Δικαστών. Η Κομισιόν θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόταση και οποιαδήποτε συνταγματική τροπολογία θα πρέπει να συζητηθεί σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την ε, σύσταση της έκθεσής σας ότι η εκλογή και η σύνθεση του Ανώτατου Συμβούλιου Εισαγγελέων και Δικαστών θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τα κριτήρια και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ένα άλλο σημείο είναι ο νέος νόμος για το διαδίκτυο που ενεκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, διότι εισάγει μια σειρά από πρόνοιες που περιορίζουν περαιτέρω την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερή, ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών. Όλες αυτές οι εξελίξεις τονίζουν το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια νέα προσέγγιση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει το σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα, έχει στρατηγικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημείο αναφοράς για τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, όπως ελέγχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Μπορεί το δυναμικό της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας να εκπληρωθεί μόνο με μια δυναμική πορεία ενταξή τη Τουρκία. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε επίσης ότι η επεξεργασία των κεφαλαίων 23 και 24 και το άνοιγμά του είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι με την προϋπόθεση ότι τα προαπαιτούμενα benchmarks ότι τα, μάλλον, ότι τα benchmarks τα οποία Έχουμε ζητήσει τα επίπεδα συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι ο βασικός άξονας των ενεργειών μεταρρύθμισης στην Τουρκία. Από αυτά που λέει η έκθεσή σας βλέπω ότι ζητάτε να υπάρξει υποστήριξη στην επανάληψη των συνομιλιών για την πλήρη λύση του κυπριακού προβλήματος και προφανώς και εμείς ως Κομισιόν χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση των ηγετών να υπογράψουν το κοινό ανακοινωθέστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρόιτε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα καταρχήν να πω το εξή. Θα ξεκινήσω από τις τελευταίες παρατηρήσεις. Κύριε Φιλόρη, αυτή η νέα νομοθεσία σχετικά με την εκλογή του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων. Αυτή η πρόταση αποσύρθηκε από το Κοινοβούλιο και αυτή τη στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις ε, με την αντιπολίτευση γιατί στόχος είναι να κατατεθεί μια νέα πρόταση και νομίζω ότι σωστό είναι αυτό. Κατ' ουσίαν αυτό είναι και το ε, αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων των Ευρωπαίων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι και εγώ ε, χαίρομαι για την δήλωση των ανακοινωθέν που υπογράφηκε σχετικά με την Κύπρο. Δηλαδή ελπίζω οι διαπραγματεύσεις ε, να οδηγήσουν ε, γρήγορα σε αίσιο τέλος. Κατόπιν, Κύριε Σοφοκλέους, απευθύνομαι σε εσά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να διαβάσετε προσεκτικά την έκθεσή μου. Κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα περιγράφονται στην έκθεσή μου. Ίσως όχι με τη διατύπωση που θα επιθυμούσατε, αλλά αναφέρομαι, ας πούμε, στις διώξεις ε, των Κούρδων. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ε, μάλλον θα σας διέφυγε ότι πέρυσι το Σεπτέμβρη ξεκίνησε μια διαδικασία Δηλαδή τώρα πλέον καταβάλλονται προσπάθειες ε, να αποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα οι Κούρδοι στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή και αν θέλετε μπορώ να σας ε, δώσω και τα σχετικά έγγραφα. Ε, αυτή τη στιγμή στόχος είναι να κατατεθούν ένα ή περισσότερα νομοσχέδια, όπως σας είπα, με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση των Κούρδων. Άρα αυτό που είπατε δεν ισχύει. Τώρα, κυρία Γιαννάκου, απευθύνομαι σε εσά Πράγματι, σε κάποια σημεία υπάρχει οπισθοχώρηση. Αν δούμε, παραδείγματο χάρη, το θέμα τη ε, δικαιοσύνη, τη ε, δικαστική εξουσία, τα μέσα ενημέρωση, τη ε, ελευθεροτυπίας και νομίζω ότι τοποθετήθηκα επ' αυτού στις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις. Εσείς ε, είπατε, όπως και οι συνάδελφοι από την Κύπρο, ότι δεν πρέπει να ανοίξουν νέα κεφάλαια. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα κεφάλαια 23 και 24 για τη δικαιοσύνη, παρόλα αυτά να ανοίξουν, γιατί αυτό είναι το αποκαλούμενο benchmark για την Τουρκία, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Πάνω σε αυτά θα μπορεί να προσανατολιστεί η Τουρκία να τα λάβει ως σημεία αναφοράς και να τοποθετηθεί στην κριτική που ασκούμε. Τάνοκ, Άτκινς και συνάδελφος Βαν Όρντεν. Ε, απευθύνομαι σε εσά, σε τρία μέλη από την ίδια πολιτική ομάδα. Ο διαπραγματεύεται για σας, για όλους. Εγώ λαμβάνω υπόψη μου τις ε, τροπολογίες σας, όμως ε, πρέπει να σας πω, έχω κατά που είπε ο κύριος Βαν Όρντεν και νομίζω ότι και ο κύριος Άτκινς έκανε μια πολύ συμπαθητική παρατήρηση όταν είπε ότι δεν του αρέσουν αυτά που κάνει το κόμμα ΚΑΠΕ. Διαπίστωσα, εν πάση περιπτώσει, ότι η Τουρκία επιθυμεί, εξακολουθεί να επιθυμεί να γίνει μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί έφυγαν από το ΕΛΚ και ε, εντάσσονται σε ένα σχηματισμό όπου πάρα πολλοί επιθυμούν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν τούτου αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας τους ανθρώπους στη δική σας την πολιτική οικογένεια. Ε, βέβαια ο τρόπος με τον οποίο ε, το παρουσιάζεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνάλφε Τάνοκ, όσον αφορά την 148 δεν συμφωνώ διότι αν και οποτεδήποτε συζητάμε για τους Αρμένιους στο Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και είμαστε προσεκτικοί. Η ε, σύνεση ε, από τότε που ήμουν εγώ εισηγήτρια οδήγησε στο ότι πολλά θέματα που παλαιότερα δεν συζητούν το καν τώρα πλέον συζητούνται και μάλιστα ανοιχτά. Δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι, αυτό είναι λάθος. Έχει αλλάξει νοτροπία σε πάρα πολλά θέματα και το ίδιο λέω απευθυνόμενοι και προς τον Αλεξάνδρ. Ε, στην παράφανεα αναφέρεται το πάρκο Γκίζη και όπου μου δίνεται ευκαιρία το κάνω. Γίνεται και αλλού στην έκθεσή μου, διότι η ελευθερία διαδηλώσεων είναι ένα ύψιστο αγαθό και νομίζω πράγματι ότι θα πρέπει να το διαδώσουμε περαιτέρω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αξίες και αυτές οι αξίες είναι κατοχυρωμένες στα κριτήρια της Κοπενχάγης. Τη στιγμή λοιπόν που μια χώρα επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και καλείται να σέβεται αυτές τις αρχές. Το λέω άρα, ίσως όχι με τη διατύπωση που επιθυμείτε εσείς Αλεξάνδρα, αλλά παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι επί της ουσίας συμφωνούμε. Συνάδελφε Τάνοκ, την 158 δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Κατόπιν, όσον αφορά τις ε, θρησκευτικές ομολογίες, τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό έγινε παράλληλα με το άνοιγμα προς τους ε, Κούρδους. Τότε λοιπόν ε, πρέπει να σας πω ότι κάτι άλλαξε για τις θρησκευτικέ ομολογίες. Έχουν περισσότερες ελευθερίες. Νομίζω ότι στον τομέα αυτό κάτι κινείται. Βεβαίως και πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα, με παρακαλέσατε γι' αυτό, αλλά Εμένα ε, με απασχολεί περισσότερο το θέμα των αλεβιτών γιατί εκεί έχω την αντίποση ότι δεν γίνονται αρκετά. Κυρία Τιεχάουζ, προσπαθώ να λάβω υπόψη μου ε, αυτά που είπατε στο βαθμό που μπορώ Κυρία Θεοχάρους, με συγχωρείτε, κυρία Θεοχάρους, ε, ίσως ε, δεν το κάνω όπως θα το θέλετε, αλλά αν δείτε επί σε τη συγκεκριμένη τροπολογία πρέπει να σας πω ότι είμαστε πολύ κοντά. Ε, πρέπει να σας πω ότι υποστηρίζω όλα αυτά που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να επιτύχουμε την επανένωση της Κύπρου. Και αναφέρω τα μεμονωμένα στοιχεία, ίσως όχι με τα δικά σας λόγια, όπως ακριβώς θα τα επιθυμούσατε, αλλά ξέρετε όταν ε, θέλει κανείς ως ηγήτρια να περάσει μια έκθεση στο κοινοβούλιο, είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει την πεπατημένη. Κυρία Λιπτσέβα, έχω ήδη μιλήσει μαζί σας ε, πριν από τη σύνταξη της έκθεσης και σας παραπέμπω στο ε, εκτιμώντας 16, εκεί ακριβώς αναφέρονται οι ανησυχίες σας. Και το ίδιο θα ήθελα να πω απευθυνόμενοι στον κύριο Χατζηγεωργίου. Ε, μου είναι απόλυτα σαφές ότι τα κεφάλαια 23 και 24 για την Κύπρο θα μπλοκαριστούν, αλλά θεωρώ ότι ειδικά τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή όπου ασκείται πίεση για θέματα δικαιοσύνης και διάκρισης εξουσιών, νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό και μέσα στην έκθεση και εκτός της έκθεσης. Αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου και αμερόληπτη δικαιοσύνη, τότε δεν είναι δυνατόν και να αντιμετωπίσει κανείς αποτελεσματικά τη διαφθορά. Η ε, κυβερνητική εξουσία δεν μπορεί να επηρεάζει ούτε το διορισμό των δικαστών, ούτε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει δικαστική ε, εξουσία αμερόληπτη. Η Τουρκία όμως πρέπει να πάρει κάποια σημεία αναφοράς, κάποια benchmarks για να γνωρίζει ε, πώς ακριβώς πρέπει να ευθυγραμμιστεί, ποια είναι τα κριτήρια, τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει νομικά και όλα αυτά να τα πράξει σε συμφωνία και σε συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας. Όλα αυτά, αυτά δηλαδή που αναφέρατε τους ε, προβληματισμούς σας, τα έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου. Ίσως να τα διατυπώνω λίγα διαφορετικά από ό,τι θα επιθυμούσατε. Πάντως νομίζω ότι το πνεύμα το δικό μου ε, ταυτίζεται με την έκθεση που εγκρίναμε πέρσι. Κύριε Σαλαβράκο, απευθύνομαι σε εσά. Πραγματικά ανησυχούμε σχετικά με την ελευθερία μέσων ενημέρωση και τύπου στην Τουρκία. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο ε, προβλέπω κάποιε συγκεκριμένε παραγράφου στην έκθεσή μου. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Σωστά ε, αυτά που είπατε τα επισημάνατε και τα συνδέσατε με το άνοιγμα του κεφαλαίου υπαριθμών 15. Προφανώς ε, δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το κεφάλαιο 15 αν δεν υπάρξει επικύρωση κάποιων ρητρών. Ε, το κεφάλαιο 15 όμως έχει και σχέση με την Κύπρο και είναι προς όφελος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Τουρκίας το να συμφωνήσουμε στο θέμα αυτό. Όμως το, η τεράστια, η πιο σημαντική προϋπόθεση το δίκαιο της θάλασσας, το UNCLOS. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι πολίτες οι καλύτες ε, πράγματι ε, επιθυμούν η Αγία Σοφία να λειτουργήσει και πάλι ως εκκλησία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ε, εγώ έχω άποψη από αυτού, αλλά δεν μπορώ να τοποθετηθώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλεξάνδρε, σας ευχαριστώ πολύ ε, για το, τη φιλοφρόνησή σας. Ε, θα θέλατε να γίνετε περισσότερο αναφορά στο Πάρκο Γκίζη. νομίζω ότι μπορείτε να δείτε λιγάκι την τροπολογία υπαριθμών 9. Και όσον αφορά το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, θέλω να σας πω ότι αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4. Εκεί γίνεται λόγος ε, και για τους ε, συμβιβασμούς. Ίσως θα πρέπει λιγάκι να είμαι πιο αυστηρή για την νομοθεσία περί διαδικτύου ενεκρίτη μόλις ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Το είπα όμως ξεκινώντας την παρέμβασή μου ότι εκεί επιθυμούμε να υπάρξει κάποια αλλαγή. Όσον αφορά την περίπτωση Γκιουλέν, εγώ θέλω να σας πω ότι κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια ε, να λάβω υπόψη μου τις σχετικές ε, τροπολογίες. Για μας, ε, για το Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόβλημα δεν είναι ο Γκουλέν, αλλά οι τουρκικές αρχές. Δηλαδή όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες και στην Τουρκία και στο εξωτερικό, στην Φιλαδέλφια τοποθετούνται επί των διαφόρων θεμάτων. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με την ε, παράκληση να αναθεωρηθούν ενδεχομένως οι τροπολογίες ε, για τον Γκουλέν. Εμείς ε, διαπραγματευόμεθα με τις αρχές και με κανέναν άλλο. Στον συνάδελφο Οπιόλτς. Νομίζω ότι ε, για τα σημαντικότερα θέματα είμαστε σύμφωνοι, για τα κρίσιμα κυρίως. Ε, θα καταλήξουμε σε καλές ε, συμβαστικές προτάσεις και νομίζω ότι η συγγήτρια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις που εκφράζονται στο Κοινοβούλιο. Καταλήγω λοιπόν, κοιτάξτε, ίσως να μην χρησιμοποιώ ακριβώς τα δικά σας λόγια, αλλά ξέρετε δεν έχει κανένα νόημα να δεχτούμε ένα σωρό τροπολογίες. Νομίζω πρέπει να είναι απόλυτα σαφές όχι μόνο λόγω της επανέναρξης διαπραγματεύσεων για την Κύπρο, αλλά και λόγω της ιδιαίτερα ευαίσθητης πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία, Νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η έκθεση αυτή να περάσει με τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία. Η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούμε να διαπραγματευόμεθα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα και παρά τα ωραία ή λιγότερο ωραία λόγια σε κάποια κράτη-μέλη καταλήγω στο συμπέρασμα ότι κανείς ε, δεν ζήτησε να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ως ε, εισηγήτρια και ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις, στην κατάσταση και για αυτό το λόγο ελπίζω ότι την έκθεσή μου θα τη στηρίξουν όλοι οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Περνάμε τώρα στην ε, έκθεση, στην σύσταση προς το Συμβούλιο της ε, κυρίας Όιουλαντ σε σχέση με τους περιορισμούς προξενικών θεωρήσεων για τους Ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Σεργέη Μαγνίτσκι. Έχετε το λόγο κυρία Όιουλαντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι γνωρίζετε την περίπτωση αυτή. Έχουμε την ε, πρότασή μας σύστασης προς το Συμβούλιο. Έχουμε αντιμετωπίσει ήδη το θέμα αυτό πριν από δύο χρόνια και ενεκρίναμε τότε το 2012, τον Οκτώβριο του 2012, την πρώτη σύσταση προς το Συμβούλιο προτείνοντας να εισαχθεί μια σειρά περιορισμών για τις προξενικές θεωρήσεις. Κυρία Όγιουλαν, συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους, αν θέλουν να φύγουν, να το κάνουν αλλά σιωπηρά, γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Όγιουλαντ, έχετε πάλι το λόγο. Φεύγουν κάποιοι, διαφεύγουν, ξεφεύγουν. Θέλουν να αποχωρήσουν από τη συζήτηση αυτού του θέματος. Όπως σας είπα, επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό ήδη για αρκετό χρόνο, παρά τις προσπαθίες μας, παρά την σύσταση που είχαμε εγκρίνει ήδη τον Οκτώβριο του 12 παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε τις αιτήσει μας με, σε διαφορετικές ευκαιρίες στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, που εμφανίζονται σε όλα τα ψηφίσματά μας για τη Ρωσία ουσιαστικά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής <clears throat> δεν έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, δεν το έχει θέσει στην ημερησία διαταξή του. Η κυρία Άστον δεν έχει θέσει το ερώτημα αυτό στο, στην ημερησία διαταξή του Συμβουλίου και φυσικά δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση από τα κράτη-μέλη. Όχι απόφαση, ούτε καν δεν έχει γίνει συζήτηση για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θέλουμε να προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναλάβει και πάλι αυτό το αίτημα και να διατυπώσει και εκ νέου αυτή τη σύσταση προς το Συμβούλιο. Προτείνουμε λοιπόν το Κοινοβούλιο να εγκρίνει μια νέα σύσταση προς το Συμβούλιο βάσει της οποίας θα επαναλάβουμε αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει ήδη στο παρελθόν του 2012 και επιπλέον αυτών των αιτήσεων ζητάμε το, Κοινοβούλιο να εγκρίνει ένα κατάλογο ατόμων για τα οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν κυρώσεις ο κατάλογος αυτός έχει εν μέρη προέλθει και από το κατάλογο του Αμερικανικού Κογκρέσου. Το Δεκέμβριο του 2012 ενέκρινε ένα νόμο για την υπόθεση Μακνίσκη το Αμερικανικό Κογκρέσο, αλλά έχουν προσθεθεί και επιπλέον ονόματα από τις διάφορες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μετά από την έγκριση της νομοθεσίας στο Αμερικανικό Κογκρέσο τα άτομα λοιπόν τα οποία κατανομάζονται στον κατάλογο αυτό κατανομάζονται βάσει μιας σαφούς τεκμηρίωσης ότι έχουν πράγματι συμπράξει στην ε, δολοφονία του Σέργεϊ Μαγνίσκι έχουν ε, ε, αρνηθεί ή έχουν αρνηθεί να του δώσουν ιατρική βοήθεια έχουν καταγραφεί ως συμμετέχοντες στην, στον βασανισμό του και στη συγκάλυψη της υπόθεσης Μαγνίσκη και επίσης έχουν συμμετάσχει στην μεταθανάτια καταδίκη του. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της σύστασης ο κατάλογος αυτός την κάνει ιδιαίτερα συγκεκριμένη τη σύσταση αυτή και την και στο Συμβούλιο μια σαφή ιδέα για το ποιοι πρέπει να είναι το αντικείμενο των κυρώσεων που θέλουμε να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζητούμε ως Κοινοβούλιο. Ο κατάλογος αυτός δεν πρέπει να θεωρηθεί ένας κλειστός κατάλογος, ένας οριστικός κατάλογος, αλλά εναπόκειται και στο Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στην πρότασή μας, να τον αναθεωρήσει, να προσθέσει ονόματα, να αφαιρέσει ονόματα εάν το θεωρεί απαραίτητο. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να παραμένει πιστό στις θέσεις που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν το 2012 συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Προτασίεβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ότι το κόμμα του ΕΛΚ έχει ζητήσει διευκρινήσει σε σχέση με την υπόθεση αυτή, την υπόθεση Μαγνίτσικη. Και έχει ζητήσει να τιμωρηθούν οι υπέτειοι στην περίπτωση μαγνηση και νομίζουμε ότι αυτή η <clears throat> πρωτοβουλία για να εγκριθεί μια σύσταση σε αυτή τη θητεία που παρουσιάστηκε από την κυρία Όγιουλαντ είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα ορθό και γι' αυτό υποστηρίζουμε απόλυτα αυτή την πρωτοβουλία και εξάλλου από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι είναι πολύ σωστό το ότι υπάρχει ένας κατάλογος υπάρχει ένας αριθμός ατόμων για τα οποία δεν έχουμε την παραμικρή ε, αμφιβολία ότι έχουν συμπράξει σε αυτή την περίπτωση. Ο κύριος Κυρίλοφ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, του Λιμπεράτκη, του ε, σκιώδους μας, πρέπει να πω ότι τούτη εδώ ε, η σύσταση αποτελεί μια πολύ καλή βάση για συζήτηση γιατί είδαμε ότι υπάρχουν ε, εξελίξεις ε, οι οποίες ε, είναι ιδιαίτερος ανησυχητικές σχετικά και όλες με το πώς φέρεται το κράτος σε αυτούς που καταδικάζουν κάποιες πράξεις και τις κάνουν δημόσιες. Ευχαριστώ κύριο Σούλτς. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ε, πολιτικής μου ομάδας θέλω να υπογραμμίσω ότι εμείς στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την έκθεση της εγκύτριας και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι αυτή η εγκληματική ιστορία σέρνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και η Κομισιόν δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Στη Ρωσία λοιπόν η περίπτωση αυτή ε, έχει, όπως σας είπα, παραταθεί, τίποτα δεν έχει γίνει και τώρα εκ των υστέρων γίνεται κάποια μεταθανάτια καταδίκη. Αυτά όλα είναι απίστευτα και θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε τον κατάλογο με την έννοια ότι τις αιτιάσεις και τις κατηγορίες για τα συγκεκριμένα άτομα να τις συμπεριλάβουμε, να ξέρουμε γιατί δεν μπορούν να εισέλθουν στη Ρουσία όσο εν περιπτώσει εξετάζεται η υπόθεση αυτή και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δοθεί ένα μήνυμα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νύχια και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για αυτούς που είναι υπεύθυνοι για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω λοιπόν και σε σχέση με την Ουκρανία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλά. Γιατί από ό,τι ακούω μέχρι τώρα η ε, ρωσική εξουσία παρισφρεί, διεισδύει στην ε, Ουκρανία, ε, παρεμβαίνει σε αυτές τις εξελίξεις με δικές της μυστικές δυνάμεις στην, στην πλατεία Μαϊντάν και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλά. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Όιλαντ και θέλω να πω και το εξής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την εντυπωσιακή και άοκνη ε, δουλειά εκ μέρους του Σεργέη Μαγνίσκη, ο οποίος αναζητούσε δικαιοσύνη ο Βίλιαμ Μπράουντον από την δική μου την εκλογική ε, περιφέρεια θέλει να, να δικαιώνεται ο Σεργέη. Και βεβαίως η δική μου πολιτική ομάδα ανησυχεί για το κράτος δικαίου και για το κλίμα αυτό ατιμορρησίας που υπάρχει στη Ρωσία. Ατιμορρησία από τη δικαιοσύνη, από αυτούς ε, που θέλησαν να ε, χαρακτηρίσουν την υπόθεση αυτή ως ε, υπόθεση ενός ε, μάρτυρος, καταγγέλλοντος μάρτυρος, έστω και εκ των υστέρων, θεωρώ ότι μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη και διαρωτώ με γιατί προσπάθησε ένας ε, ε, Ρώσος διπλωμάτης να το δικαιολογήσει ότι μπορεί κανείς ε, να διώκει και μετά θάνατον κατηγορούμενους. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις σε όσους είναι υπεύθυνοι. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το Αμερικανικό Κογκρέσο και άλλοι πολλοί έχουν δεσμευτεί για αυτή την υπόθεση Βεβαίως δεν είμαστε απόλυτα αρμόδιοι για το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι η θέση που θα λάβει το δικό μας το Κοινοβούλιο είναι ένα μήνυμα που εκπέμπεται και θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την επιμονή που δείχνει στο να αντιμετωπίσει σχετικά με αυτή την υπόθεση. Και υπάρχει μία παράγραφος όμως ε, στο σχέδιο του κειμένου που θέλω να υπογραμμίσω, εκεί όπου γίνεται λόγος ότι είναι ε, όλο και περισσότερο απαραίτητο να ε, εξεταστεί η κατάσταση στη Ρωσία. Γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε. Μέχρι τώρα οι παραβιάσεις της Ρωσίας στις διεθνείς της δεσμεύσεις είναι εντυπωσιακέ. Όσο λοιπόν συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε ότι ανησυχούμε, ότι ε, δεν συμφωνούμε. Βλέπουμε αυτό δεν αρκεί σε μια πολιτικά διεφθαρμένη κοινωνία τα συγκεκριμένα στοχευμένα μέσα, μόνο αυτά μπορούν να επιφέρουν ε, αποτέλεσμα. Και η υπόθεση Μακνίτσκι είναι καλά τεκμηριωμένη, γι' αυτό λοιπόν όπως και το Κογκρέσιο των ΗΠΑ θα πρέπει και εμείς να καταρτήσουμε έναν κατάλογο ατόμων που ευθύνονται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετίζονται με το θάνατο του κυρίου Μαγνίτσκι. Ίσως μπορούμε και το απόγευμα να ρωτήσουμε την ύπατη εκπρόσωπο γιατί δεν κατόρθωσε το θέμα αυτό να το συμπεριλάβει στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα εχθές. Ο κύριος Λαντσμπέρκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται για την περίπτωση και μονάχα. Είναι και θέμα συνεκτικότητας και αξιοπρέπειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή μας και ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραμείνει σαφής και προσιλωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην προσπαθεί <clears throat> να καλοπιάσει κατά κάποιο τρόπο δικτατορικά καθεστώτα θα πρέπει να καταγγείλει όλους τους δολοφόνους και βασανιστές. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτή την, αυτή την πρωτοβουλία της Κριστίνα Όγιουλαντ, η οποία είναι απόλυτα ορθή. Ευχαριστώ πολύ. Από την ε, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων DG Home της Κομισιόν, η κυρία Σμιτ και ο κύριος Πάλμεν θα λάβουν το λόγο και θα μας εξηγήσουν ποια είναι η δική τους θέση σε σχέση με την άποψη του, της Επιτροπής μας. Κυρία Σμιτ. Κύριε Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Dietrich Πάλμεν από τη Γενική Διεύθυνση Home, DG Home. Η πρώτη μας αντίδραση θα πρέπει να προέλθει από την, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί αυτό δεν εμπίπτει στις δικές μας αρμοδιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να δώσετε το λόγο στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τα έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι εφιστούν την προσοχή μας στην περίπτωση Μαγνίτσκι. Δυστυχώς δεν είναι μοναδική αυτή η περίπτωση, όπως ελέγχθη, είναι μια περίπτωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ρωσία. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις με την πλήρη προσοχή που απαιτούν, γιατί βλέποντας αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να υπογραμμίσουμε τα συστημικά προβλήματα και τις αστοχίες που υπάρχουν στην προφυλάκηση, όπως την περίπτωση της κ. Νικολίκοβα, τις ε, συνθήκες κράτησης που είναι πάρα πολύ δυσμενείς και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με όλα αυτά τα δικαστικά προβλήματα και εμείς φυσικά υποστηρίζουμε όλους τους ακτιβιστές οι οποίοι εμπλέκονται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα και χάρη στη βοήθεια του Κοινοβουλίου έχουμε δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ για τους ακτιβιστές αυτούς. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, Παρακολου... ερχόμαστε σε επαφή με τις οικογένειες, τους ε, δικηγόρους του κ. Μαγνίτσκι και με όλους τους εμπλεκόμενους για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει σε σχέση με αυτά τα θέματα. Για την περίπτωση Μαγνίτσκι έχουν ελεχθεί τα πάντα από τους ε, κύριους βουλευτές είναι εδώ σαφές ότι έχει αποτύχει ο αγώνας κατά της διαφθοράς και επίσης έχει αστοχήσει το δικαστικό σύστημα. Έγιναν έρευνες από ανεξάρτητους φορείς στη Ρωσία, όπως το Συμβούλιο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων του Πρόεδρου της Ρωσίας, που κατέληξαν και το Συμβούλιο για τις ε, Φυλακές που κατέδειξαν ότι πραγματικά υπήρξαν σημαντικές ελλείψεις και ενοχές για τα θέματα αυτά και περιμένουμε <clears throat> και όλες αυτές οι εκθέσεις συνάδουν με τα συμπεράσματα αυτά που αναφέρετε και εσείς. Τι μπορεί να γίνει τώρα παραπάνω. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Πρώτα απ' όλα είναι κάπως μοναδική η κατάσταση όταν ο, κύριος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέστειλε μια επιστολή για το θέμα αυτό στον ε, τότε ομόλογο του κύριο Μετβέντεφ για την περίπτωση Μετβέντεφ, για την Μαγνίσκη, συγγνώμη, ζητώντας οι ρωσικές αρχές να κάνουν τις απαραίτητες έρευνες. Οι προσπάθειες λοιπόν του Συμβουλίου και της κυρίας Άστον που έχει εκδώσει δύο δηλώσεις για την περίπτωση Μαγνίσκη δείχνουν την προσοχή που έχουμε δώσει. Ακόμα και αν το θέμα αυτό λοιπόν δεν ήταν στη μέση διαδράξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, σίγουρα είναι στις οθόνες μας και παρακολουθούμε το θέμα αυτό με κάθε προσοχή. Εγώ προεδρεύω των ε, συναντήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη Ρωσία και το θέμα αυτό επανέρχεται στις συζητήσεις μας. Καταλαβαίνω η ματέωση που νιώθετε γιατί η απάντηση των ρωσικών αρχών για τα θέματα αυτά είναι ότι εμείς πολιτικοποιούμε μια υπόθεση της ρωσικής δικαιοσύνης και αυτή είναι η μόνη απάντηση που μας δίνουν. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε. όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης που υπογραμμίζει την ε, ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε την ε, απαγόρευση προξενικών θεωρήσεων και το πάγωμα των καταθέσεων στο εξωτερικό σαν μια τελική λύση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό φυσικά δεν αποκλείεται να γίνει, αλλά αν το κάνουμε θα πρέπει να δούμε τι συνέπειες θα προκύψουν και οι συναδελφοί μου μπορούν να σας υπογραμμίσουν τι θα προκύψει. Είναι σαφές ότι έχουμε κάποιες εμπειρίες με τις κυρώσεις και εδώ πρέπει να έχουμε την σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών, αλλά κυρίως ξέρουμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες στο παρελθόν, γιατί τα άτομα που βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορούν να πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να διαμφισβητήσουν την εγγραφή τους σε αυτή τη λίστα. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν αυτό το δρόμο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες οι οποίες μπορούν να προκύψουν και οι οποίες θα είναι φυσικά πολύ αρνητικές αν τα άτομα αυτά καταφέρουν ενώπιον των δικαστηρίων να καταδείξουν ότι δεν πρέπει να είναι στον κατάλογο αυτό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια πιο ε, βαθμιαία απάντηση σε όλα αυτά, να ζητήσουμε από τις ρωσικές αρχές να κάνουν πλήρεις έρευνες στα θέματα αυτά και σε περίπτωση που δεν υπάρξει αντίδραση από τις ε, ε, ρωσικές αρχές. Ήδη το κοινοβούλιο σας είχε ήδη κάνει κάποιες ε, ε, προτάσεις σε σχέση με τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Υποξενικών Θεωρήσεων που είναι υποδιαπραγμάτευση και αυτός είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό πρώτου περάσουμε σε πραγματικές κυρώσεις. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για την στήριξη. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, που συμπεραίνω λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ε, με την ε, σύσταση. Θα περιμένω τις τροπολογίες ε, που υποσχέθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι ότι θα υποβάλουν και θα δούμε τι δυνατότητες έχουμε ακόμα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θέλω να πω, μέχρι να τελειώσει η θητεία μας. Ευχαριστώ. Να σας πω λοιπόν ότι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 27 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Κύριε Λάντσπαρκ, σύντομα ανακοινώσατε τροποποιημένο ε, χρονοδιάγραμμα για την σύσταση για την Τουρκία, γιατί η Ρία κάτι είπε σχετικά, αλλά εμείς δεν ακούσαμε τις νέες ημερομηνίε. Ίσως ε, φταίω εγώ, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος. Υπάρχει λοιπόν νέο χρονοδιάγραμμα για την σύσταση για την Τουρκία ε, ή ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Γιατί σίγουρα δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Ναι, γιατί η Ιρία ζήτησε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Έτσι δεν είναι. Πρόεδρος, εδώ που βλέπω εδώ, αυτό που βλέπω εδώ γραμμένο, αλλά μάλλον ε, είναι πλέον ξεπερασμένο, λέει ότι θα ψηφιστεί η σύσταση αυτή την 3η Μαρτίου. Όχι, αλλά διαβάζω λάθος γιατί μία αναφέρεται στο 13, εμείς είμαστε 14 τώρα. Ναι, τώρα αυτό έχω εγώ γραμμένο. Okay, we'll have a break. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι την έναρξη του διαβριμένου Προεδρείου όταν θα έρθουν, όταν θα έρθουν πλέον όσοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν εις το διευρυμένο Προεδρείο. Τα λέμε σε λίγο.